Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη έναρξη της ε, συνεδρίασής μας, αλλά οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι όπως γνωρίζετε και επομένως έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα πρόσβαση στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα σας πω ότι συζητήσαμε στους ε, συντονιστές στη συνεδρίαση που είχαμε χτες το βράδυ. Διορισμός εισηγητών για την ενόψη των εκλογών του 2014, και Γουελτιέρη είναι οι Όσον αφορά τη γνωμοδότηση για τις στατιστικές, ε, ο υποφαινόμενος, ο πρόεδρος σας ε, θα συντάξει γνωμοδότηση. Η, η ψηφοφορία η οποία είχε προβλεφθεί για σήμερα το πρωί ε, όμως αφαιρέθηκε γιατί ε, γιατί δυστυχώς και εγώ δεν θα είμαι διαρκώς εδώ. Έχω κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσω και δεν θα είμαι δυστυχώς συνέχεια εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ο εισηγητής αρμόδιας επιτροπής θα ε, μας ε, ζητήσει, θα μας πει πότε θα γίνει η τελική ε, συζήτηση και ψηφοφορία. Επίσης, ε, πρόταση πρωτοβουλίας ε, της Γιούρη όσον αφορά τον έλεγχο των εξουσιών της Κομισιόν. Ο εισηγητής θα βρίσκεται την επόμενη συνεδρίαση. Ένα νέο σχέδιο εκθεσής θα υποβληθεί από τον συνάδελφο Νταφ όσον αφορά το πρωτόκολλο της Τσεχικής Δημοκρατίας. έχει ζητηθεί η ερμηνεία του άρθρου 159, αλλά οι συντονιστές ε, ε, πρότειναν πριν ε, εκφραστούμε εμείς να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία και ούτως θα πράξουμε. επίση θα κάνουμε και έκθεση για την τροποποίηση 7 του, κανονισμού, για του άρθρου 7 του κανονισμού όσον αφορά την περίπτωση άρσης ημί της ε, ασυλίας ε, σε ε, περιπτώσεις που υφίσταται συνέχεια από προηγούμενες αποφάσεις. Επίσης, συνεδριάσει βάσει του άρθρου 51 όσον αφορά το πρόγραμμα της ε, για το οποίο έχει ήδη προβληθεί η εφαρμογή του ιδίου άρθρου 59. Ξέρετε ότι ε, η Επιτροπή Γιούρη είχε συζητήσει το θέμα αυτό. Τον Φεβρουάριο του 2013 θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να γίνει σεμινάριο ε, με δύο θέματα το πρωί ε, μετά από αίτημα του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας θα έχουμε διάσκεψη με συμμετοχή ε, των εκπροσώπων των ε, Ιδρυμάτων με θέμα ε, πολιτικά Ιδρύματα στην Ευρώπη, πέντε χρόνια πολιτικής πρόθεσης. Το απόγευμα θα, το θέμα θα είναι η πρόσβαση στην ψήφο, δικαίωμα ψήφου σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές εκλογές και ευρωπαϊκές εκλογές επίσης. Πρόκειται για ένα θέμα ε, πρόσβαση στην ψήφο και ηθαγένεια. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας έχει ε, αποσχολήσει ε, ήδη πριν από λίγο χρόνο. Αυτά ήθελα να σας πω και μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε με την ίδια διάταξη, σημείο 11 εξέταση προβλημάτων συνταγματική φύση από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνησυγητέ είναι οι ε, Τσαρκόφσκι και Γκουαλτιέρη. Έχουμε συζητήσει μια πρώτη φορά το θέμα, δεν έχουμε έγγραφο εργασία. Ελπίζω συντόμω να το έχουμε. Θα ακούσουμε πάντως πρώτα τους δύο συνεισηγητές. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτα, ο συνάδελφος Τσαρκόφσκι ή ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη. Ο Ταρκόφσκι, εντάξει, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Έχω μια καλή ενακτήρια φράση. Εργαζόμαστε για το έγγραφο εργασίας. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουμε εξάλλου. Βρισκόμαστε στην ορθή κατεύθυνση και πορεία. Διότι θεσπίσαμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε πάνω κάτω και έχουμε και τους ορισμούς όσον αφορά την πολυδιακυβέρνηση, πολυδιαχείριση για την αποσαφήνιση θεμάτων και όπως είχαμε πει και προηγούμενα, σε άλλες συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Πρώτα θέλουμε να συζητήσουμε για την κινητοποίηση του δυναμικού της υφιστάμενης συνθήκης, της κείμενης συνθήκης. Τι μπορεί να γίνει και τι είναι εφικτό υπό το πλαίσιο των συνθήκων ως έχουν. Και αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο, διότι ουσιαστικά η συζήτηση διεξάγεται για το ίμιου, αλλά όχι μόνο για αυτό, αλλά υπάρχει και το τι μπορούμε να κάνουμε δεδομένων των προϋποθέσεων υπό τις οποίες εργαζόμαστε. Βλέποντας στο μέλλον τι θα ήταν δυνατόν και εφικτό αν μπορούσαν να αλλάξουν οι συνθήκες και τις προσαρμόζαμε. Και εξειδικευμένα προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η ευρωδιακυβέρνηση χρησιμοποιώντας το μέγιστο τις συγκεκριμένες δυνατότητες που προσφέρουν οι συνθήκες και όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές, την πολιτική για την απασχόληση, και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπου εργαζόμαστε ακριβώς στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή προετοιμάζοντας ακριβώς γνωμοδοτήσεις νομιμότητα θεμητό των εργασιών μας, διαφάνεια ευρωπαϊκό εξάμεινο, εποπτεία τραπεζών, όλα αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση και συζήτηση στο πλαίσιο της βελτίωσης της ε, Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης προσπαθώντας να στραφούμε και στο μέλλον να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον προβλέποντας και εξετάζοντας δυνατότητες για την ε, ε, Δημοσιονομική Ένωση και ίσως Πολιτική Ένωση κάποια μέρα. Και τέλος τέλος αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι προσπαθούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στις μελλοντικές ε, αλλαγές στις συνθήκες και να δούμε την προοπτική στο μέλλον πώς θα μπορούσαν αυτές οι αλλαγές, οι προσαρμογές να συμπληρώνουν τα όσα κάνουμε τώρα και να δούμε την προοπτική συνέχεια αυτών στο μέλλον και να δούμε πώς μπορούν να εξεταστούν αυτές οι δυνατότητες αλλαγή συνθήκων. Το πιο σημαντικό είναι φυσικά το να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ιδέες, υπογραμμίζοντας αυτές, αυτό είναι το νόημα αυτού του εγχειρήματος, τονίζοντας και παρουσιάζοντας αυτά που επιθυμούμε. Όλα αυτά που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παρεμβάσεις, αλλά επίσης και αυτά τα οποία επιβεβαιώθηκαν μετά από ακροάσεις που κάναμε πιο σημαντικό, πιο σημαντικά από αυτά, να εμβαθύνουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, βασιζόμενη πάντα στις μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα, χωρίς να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, χωρίς να περάσουμε σε διακυβερνητική μεθοδολογία ή προσέγγιση. Προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε και να πούμε ότι σε σχέση με αυτήν την παλαιά διαφοροποίηση που έχει καταστεί ανεδαφική πλέον, κάνουμε λόγο και για τον κατακαιρματισμό όσων το γίνονται για το επίπεδο πολυδιακυβέρνησης που θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες διαφορές. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να τεθούν προτεραιότητες για το μέλλον, αλλά επίσης και να πούμε με σαφήνεια ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτής της Ευρωβουλής. Τι έχει υπόψη η Ευρωβουλή να κάνει και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Να οικοδομήσουμε σε αυτά που επετεύχθησαν ως θεμέλια από τους οδηγούς Σέρπας, οι συντονιστές κατά το παρελθόν και σε σχέση με διαβουλεύσεις να μπορέσουμε από αυτή την αφετηρία να προχωρήσουμε και να, ε, να δομήσουμε κάτι. Επί ποιου θέματος εργαζόμαστε τώρα. Εξετάζουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε ποια συγκεκριμένα σημεία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε όλα αυτά. Και εδώ πρόβλημα υπό τη σημερινή κατάσταση όσο έχουν οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά κάποιες ιδέες θα μπορούσαν να, να αποτελούν κάποια πρόκληση. Δεν είναι απόλυτη η βεβαιότητα από πλευρά μα τι θα μπορούσε να γίνει και πρέπει να δούμε και σε σχέση με την προοπτική αλλαγή συνθήκων αν θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι τι μπορεί να γίνει. Να προετοιμάσουμε έτσι προβληματιζόμενοι σε αυτό το πεδίο να δούμε αν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πείθοντας το θέμα να, να μπορέσουμε στο μέλλον να προβάλλουμε τις επιθυμίες αυτές ώστε να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε σε σχέση π.χ. και με όποιες αλλαγές χρειαστούν. Αυτά σε σχέση με τη δομή όσον αφορά την ε, έκθεση υπό Προσπαθήσαμε να, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την εξή διαδικασία. Πρώτον, να παρουσιαστεί όχι η έκθεση πρώτα, αλλά ένα έγγραφο εργασίας σε αυτή τη φάση. Θέλουμε να συζητήσουμε τη διάθεση, τη δομή μαζί σας και τις φιλοδοξίες, ε, τις προσδοκίες και τους στόχους αυτής της έκθεσης προτού διατυπωθούν τελικά αυτές οι δομές και αυτές οι προτάσεις ώστε να διαβουλευτούμε επ' αυτών και να υπάρξει μέγιστη υποστήριξη από τα μέλη των θεμάτων αυτής της έκθεσης. Ας το πω έτσι μια περίληψη εν συνόψη των φιλοδοξιών μας, των προσδοκιών μας και των στόχων μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, κύριε Ταρκόφσκι, μας ε, δώσατε ένα δίκτυ εργασίας για το παρελθόν και για το μέλλον. Ο κύριος Γκολτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσθέσω δύο λόγια σε αυτά που είπε ήδη ο Ραφέλη. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, πιστεύω ότι και η επερχόμενη τελική έκθεση ε, Φαν Ρομπόη θα πρέπει να ε, μας, ε, μάλλον να την περιμένουμε πριν προχωρήσουμε στην τελική εκδοχή της έκθεσής μας. Είχαμε και την έκθεση Tyson από μερικές μέρες. Νομίζω ότι έτσι έχουμε ακόμα περισσότερα επιχειρήματα έτσι ώστε που συνηγορούν μάλλον υπέρ της ε, αναβολής ε, της εργασίας. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής μας ε, ΑΦΚΟ και φαντάζομαι ότι το έγγραφο εργασίας θα είμαστε σε θέση να το μοιράσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. πολυεπίπεδη είπαμε θα είναι η αντιμετώπιση του θέματος. Να πω δύο λόγια γι' αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι είδους πολυεπίπεδη θα είναι αυτή η προσέγγιση so far uh, uh, uh, ε, θα δούμε λοιπόν ε, ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την πολυεπίπεδη ας πούμε διακυβέρνηση και όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης. Ξεκινάμε από την βασική από το βασικό διαχωρισμό χώρες ευρώ και χώρες μη ευρώ. Πιστεύω ότι και από πολιτική άποψη αλλά και από θεσμική αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ανάμιξη και να αναφερθούμε στις χώρες οι οποίες ε, ακολούθησαν το opting out αλλά και χώρες οι οποίες ναι μεν αυτή τη στιγμή εξαιρούνται αλλά έχουν δεσμευτεί να ε, μπουν στο ευρώ. Επίσης πιστεύω ότι ως βάση ε, για την πολυεπίπεδη αντιμετώπιση θα πρέπει ε, να πάρουμε αυτήν την, ε, αυτόν τον διαχωρισμό και να μιλήσουμε βεβαίως ε, και για τους πόρους γιατί για εκεί υπάρχει αυτή η διάκριση. Επίσης θα πρέπει να εισαχθεί το ζήτημα του Fiscal Compact. Γιατί εκεί το σχήμα είναι διαφορετικό. Έχουμε 25 χώρες. Έχουμε την Δανία ε, που είναι εντός του συμφώνου και την Τσεχία που είναι εκτός. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι λάτρης του Fiscal Compact, αλλά αυτό που είναι σημαντικό από θεσμική άποψη είναι το γεγονός ότι εγκαθιδρεί de facto ένα νέο ίδρυμα, ας πούμε, ή ένα νέο καθεστώς που είναι η διάσκεψη κορυφής, τον, ε, το Euro Summit. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μέσα από τη συζήτηση ε, τελικά διευρύνθηκε κατά κάποιο τρόπο η συζήτηση το, της Ευρωζώνης ε, συμπεριλαμβάνοντας και χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτεί να μπουν στο ευρώ αργότερα. Και βεβαίως εδώ εμπλέκεται και το Κοινοβούλιο σαν ε, σώμα, σαν ένα σώμα που έχει ισχυρό πολιτικό στίγμα. Και έχουμε βεβαίως και το Eurogroup, το οποίο παρότι δεν είναι τόσο επίσημο, κάνει πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι έχοντας αυτά τα τρία θεσμικά στοιχεία, μπορούμε να δούμε ε, το μοντέλο το οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε. Γιατί αν αναλογιστούμε το μοντέλο που εκτενώς εξηγήθηκε από την καγκελάριο Μέρκελ στο λόγο της στο Κοινοβούλιο, ε, εκείνη αναφέρεται ε, σε μια ένωση σταθερότητας και διπλής δύναμης. Ε, δεν νομίζω ότι όμως ότι θα μείνουμε εκεί, γιατί βλέποντας την ουσία καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μοντέλο μιας ένωσης κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κανόνες, αυτό είναι σαφές και νομίζω ότι πλέον οι δυνάμεις της αγοράς είναι αυτές οι οποίες θα κινήσουν τελικά την οικονομία και θα διαμορφώσουν τους ε, κανόνες. Και εμείς απλώς ε, θέλουμε να ε, βάλουμε κάποιους κανόνες σαν συγκεκριμένους κυβερνητικούς κανόνες διακυβέρνησης που θα δώσουν περισσότερη ουσία θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα είδος executive federalism. και θα ξεφύγουμε ίσως από τους κανόνες που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός πολυεπίπεδης διακυβέρνησης έτσι όπως, ε, από τη, έτσι όπως προβλέπεται από τις συνθήκες μπορεί να μας ε, οδηγήσει στο δρόμο που τελικά θα μας κάνει να φτάσουμε σε πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση. Governance ε, Επομένως, μπορούμε να δουλέψουμε καλά χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα εργαλεία. Εάν βέβαια εισαχθεί και το στοιχείο της επιπλέον δημοσιονομικής ε, ικανότητας, Εάν βάλουμε δηλαδή και το στοιχείο των πόρων και αν από πολιτική άποψη δούμε ότι δεν φαίνεται πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία στους 27 και αν αποφασίσουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την ε, δυναμωμένη δημοσιονομική ικανότητα όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα τότε μπαίνουμε σε ένα νέο χώρο και θα πρέπει να σκεφτούμε πλέον την επίδραση που θα έχει ε, ε, η εισαγωγή διαφορετικών επιπέδων που όχι μόνο θα διέπονται από διαφορετικούς κανόνες αλλά μπορούν να οδηγήσουν και σε διαφορετικούς πόρους και διαφορετική φορολογική ικανότητα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε, να τα επεξεργαστούμε στην ε, έκθεσή μας και νομίζω ότι ένα από τα αποτελέσματα δεν θα είναι να βάλουμε ένα τείχο ανάμεσα στην, ε, στις χώρες ε, της Ευρωζώνης και τις υπόλοιπες, αλλά αντίθετα να δούμε τις διαφορές ε, ανάμεσα το, ανάμεσα στις χώρες του ευρώ μαζί με τις χώρες οι οποίες έχουν επιτύχει εξαίρεση μέχρι τώρα από τη μία μεριά και τις χώρες που έχουν επιλέξει να είναι έξω από το ευρώ από την άλλη. Θα πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα ταυτοποιεί τις δυνατότητες δημιουργίας γεφυρών ε, που θα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολυεπίπεδης δημοσιονομικής ικανότητας και οπωσδήποτε θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ε, σε μοντέλα όπως είναι το ETF εκτός του προϋπολογισμού αλλά και μοντέλα εντός του προϋπολογισμού που όμως θα βασίζονται σε διαφορετική προετοιμασία και διαφορετική ε, σκοπιά. που θα βασίζονται και στην ε, πραγματικά ε, δημοσιονομική, συγγνώμη, στην πραγματική προϋπολογιστική δημοσιονομική ικανότητα κλπ. Όμως, συμφωνώ και με τον Ράφα σε αυτό, ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο, γιατί άλλωστε έχουμε και μια τέτοια εντολή στην έκθεση Tyson, ας πούμε, αναφέρεται ότι έστω και αν θεωρούμε ότι η μελλοντική συνθήκη θα καταστεί δυνατή αργότερα μετά τις εκλογές, όχι πριν από το 2015, εν πάση περιπτώσει, αλλά αναφέρεται επίσης ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τις σκέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή των συνθήκων θα μπορούσε να ενισχύσει την ε, δυνατότητα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ε, που βασίζεται όχι μονάχα σε διαφορετικούς κανόνες αλλά και σε διαφορετικούς πόρους. Πολλή δουλειά έχουμε να κάνουμε και ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι βεβαίω θα μας δώσουν ε, και ενδιαφέρουσες απόψεις τις οποίες θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στην εκπόνηση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ο συνάδελφος Νταφ έχει ζητήσει ήδη το λόγο. Μάλιστα, πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συνεισηγητάς για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή τους. Έχω όμως και δύο-τρία σχόλια. Για να καταλήξουμε σε μία θαυμάσια έκθεση, γιατί θαυμάσια πρέπει να είναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε για τη σύμβαση, για τη συνέλευση. Ξέρω ότι είναι για το 15, αλλά μέχρι τότε αποσιοποιητικά. Πρέπει να προετοιμαστούμε πριν αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία. ώστε να είμαστε πλήρως έτοιμοι. Άρα Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε ορισμένες πρώτες σκέψεις γιατί η Κομισιόν απειλεί να δημοσιεύσει εκείνη οδηγίες για τη μελλοντική ζωή της Ένωσης, κυρίως τα φορολογικά και δημοσιονομικά. Και πρέπει τουλάχιστον να συνεννοηθούμε με την Κομισιόν από σταθερή και υπεύθυνη θέση και πλήρως ενημερωμένη. Ελπίζω το Δεκέμβριο το Συμβούλιο στα συμπεράσματα μάλλον της Προεδρίας να μιλήσει και για την Πολιτική Ένωση και να δεσμευτούν οι πρωθυπουργοί για επίσημη αλλαγή της συνθήκης το 15 αλλά επίσης και ότι θα αρχίσουν, θα ζητήσουν μία προπαρασκευαστική τουλάχιστον περίοδο ανάλυσης όπου το, κατά την οποία το κοινοβούλιο να παίζει σημαντικό ρόλο. Να είναι παρόν δηλαδή. αν συμφωνηθεί τελικά να υπάρξει εμβάθυνση της πολιτικής ολοκλήρωσης. Με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα αυτά που είπε η καγκελάριος Μέρκελ της προάλλες εδώ στο κοινοβούλιο. Γιατί η προηγούμενη ομιλία της στην Βρύγη, όπου έκανε λόγο για την ενωσιακή μέθοδο μου είχε φανεί κλασική, τυπική, διακυβερνητική δήλωση, ενώ τώρα έχει αλλάξει στάση από τότε, από την ομιλία της Βρύγης. Μίλησε για τη σημασία της Κομισιόν ως εκτελεστικής αρχής και επίσης μίλησε για τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να το αναγνωρίσουμε δε αυτό επίσημα, αυτή την αλλαγή δηλαδή στην γερμανική ανάλυση και στάση, πιστεύω ότι καιρός είναι το Κοινοβούλιο επίσης να κάνει μια χειρονομία να καθησυχάσει την Ευρωζώνη, τα μέλη της Ευρωζώνης, ότι και εμείς είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα ήθη μας και να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη φύση που έχουν οι λήψεις δημοσιονομικών αποφάσεων για την Ευρωζώνη. Ίσως να μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη δημιουργία μιας Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωζώνης στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών αφήνοντας φυσικά την Ολομέλεια ως τελευταίο λόγο σε όλα τα μέλη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά για τα προπαρασκευαστική δουλειά αυτή να δίνεται να γίνεται από αυτή την ειδική υποεπιτροπή εποπτείας της Ευρωζώνης. Αυτό νομίζω πρέπει να το πείτε στην έκθεσή σας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επίπτωση των πολυεπίπεδων στη δουλειά του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, Όπως βλέπουμε και από τις εφημερίδες, τα έθνη που δεν διαθέτουν κράτος, όπως η Σκοτία, η Καταλανία, ίσως και άλλα, αρχίζουν να παίζουν σημαντικότερο ρόλο και πρέπει να αναρωτηθούμε Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την θεμητότατη εξέλιξη των εθνών χωρίς χωρίς να αλλάξουμε το ρόλο των υπαρχών των κρατών μελών ή χωρίς να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό τους. μπορούν να υπάρξουν απαντήσεις και είμαι ακόμη υπέρ της πρότασής μου για τα διεθνικά ψηφοδέλτια για το Κοινοβούλιο και τις εκλογικές περιφέρειες που να ταυτίζονται περισσότερο με τις ιστορικές όπως στην Ισπανία και στην Μπολονία. Νομίζω ότι καλό θα ήταν η έκθεσή σας επίσης να μιλάει και για αυτό το καινούριο φαινόμενο. Επίσης, θα έπρεπε ίσως να προσαρμοστεί ο ρόλος, να αλλάξει ο ρόλος των χωρών μελών ώστε να γίνει μια σαφή ρητή πρόταση για μικρότερη κομισιόν. Φυσικά στη Λισαβόνα δεν το πετύχαμε αυτό γιατί έγινε δεκτή αυτή η παράλογη ιδέα ότι οι πρωθυπουργοί θα έπρεπε λέει να βρουν έναν τρόπο να διασφαλίζουν την εκπροσώπηση των δύο τρίτων των εθνικοτήτων. Αλλά αυτό δεν γίνεται βέβαια και ανέκαθεν ήταν παράλογο να θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Την επόμενη φορά λοιπόν πρέπει ρητά να πούμε ότι ζητάμε μικρότερη κομισιόν τις οποίας τα μέλη να διορίζονται από τον πρόεδρο αλλά να εκλέγονται από το κοινοβούλιο ή μάλλον να μην διορίζονται από τον πρόεδρο αλλά να εκλέγονται από το κοινοβούλιο. Έτσι θα σπάσει ο φαύλος κύκλος σύνδεσης του Επιτρόπου με τη χώρα του που έχει μειώσει <clears throat> την ποιότητα της δουλειάς, της νομοθετικής δουλειάς. Τέταρτον, να πούμε κάτι για την στάση της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας. Και οι τρεις έχουν κάποια ασταθή και μη ικανοποιητική σχέση με την Ένωση. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί για επικοδομητική λογική ανάλυση και πολυεπίπεδη, τότε πρέπει να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να το πούμε και στη νέα συνθήκη κάτι και για τέτοιες χώρες που που σαν την Τουρκία Μπορεί να μην θελήσουν να μπουν στην Ένωση. Ή χώρες που θέλουν αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν. ή και για υπάρχουσες χώρες μέλη που δεν θέλουν να κάνουν το ομοσπονδιακό βήμα που ζητούν οι υπόλοιπες. Και πρέπει λοιπόν να βρεθεί κάποιος αξιόπιστος και βιώσιμος τρόπος σχέσης και με αυτές. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης συζήτηση της πολυπαιδικότητας αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα των χωρών αυτών. Σα ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Έχω ακόμα άλλον έναν εγγεγραμμένο, τον κύριο Μπρόντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. ερώτηση μάλλον που προκύπτει από αυτά που είπε ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη που είπε ότι η ε, πραγματική διαφοροποίηση δεν είναι μεταξύ των 17 που είναι Ευρωζώνη και των 10 που δεν είναι, αλλά ε, το, το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει ας πούμε opt-out και τους άλλους 9 που δεν έχουν. Αναρωτιέμαι. Πόσο σίγουροι είστε και εσείς και άλλοι ότι άλλοι πραγματικά θα θελήσουν να μπουν στην ε, ε, Ευρωζώνη και αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν τελικά υπάρχει κάποια δυνατότητα, κάποιος, ε, κάποιος τρόπος να, τους, να εξαναγκαστούν να μπουν στο ευρώ. Οι εννέα συν τα μελλοντικά μέλη οπωσδήποτε θα μπουν στην Ευρωζώνη και τότε το, το Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα στην πολυεπίπεδη ε, ε, διακυβέρνηση. Δεν ξέρω εάν καταλαβαίνετε τι σας ρωτάω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Είναι μια πολύ, ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό σημείο επί του οποίου πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι εμείς ως Συνταγματική Επιτροπή πρέπει περισσότερο να δούμε τις πραγματικές διεργασίες και διαδικασίες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τι γίνεται στην πραγματική ζωή, αν θέλουμε να τις προτάσεις μας για τη μελλοντική διακυβέρνηση να συμφωνήσουμε επί των προτάσεων αυτών στο μέλλον. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ουσιαστικά και με τις ρυθμίσεις για την νομισματική ολοκλήρωση από τη συνθήκη του Μαστρίχτα αν σήμερα εμεί θέλουμε να συμφωνήσουμε προς μια κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε αυτό σημαίνει ότι πρέπει επί των αρχών να σκεφτούμε πώς μια οικονομική νομισματική ένωση θα διαμορφωθεί η οποία θεωρητικά θα αποτελείται από 27 ή 28 κράτη-μέλη ή δηλαδή η 28 κρατη μελη η δηλαδη δυνατοτητα που θα δημιουργηθεί σε σχέση με την ε, συνεργασία για τα θέματα οικονομικής νομισματικής ένωσης και για την, ε, το ενιαίο νόμισμα θα πρέπει να διαβουλευτούμε και να δούμε ότι αυτή η πορεία μέσω του ενιαίου νομίσματος θα πρέπει να οδηγήσει μια, σε έναν εναρμονισμό των οικονομικών και νομισματικών συνθήκων στην Ευρώπη. Δηλαδή μέσα από το πολιτικό πλαίσιο πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πώς αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να αναδιοργανωθούν για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Συμφωνώ μαζί σας, χρειαζόμαστε μάλλον αλλαγή των συνθήκων, μια συνταγματική ε, διακυβερνητική διάσκεψη και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς θα εκδημοκρατικοποιήσουμε όλο αυτό το οικοδόμημα. Και φτάνω σε δύο σημεία που θέλω να αναφέρω. Δεν ξέρω αν τόσο απλά έναντι της πραγματικότητας μπορούμε να προσαρμοστούμε και να ακολουθήσουμε κάποιες τάσεις. Έχουμε την Ευρωζώνη. Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη σε σχέση με ισοδίκια και ισότιμη συμμετοχή που θα πρέπει να διασφαλίζεται για τις αποφάσεις για την προοπτική αυτής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όταν λέμε το ενιαίο νόμισμα χρειάζεται μια ενιαία οικονομική πολιτική, μια ενιαία δημοσιονομική πολιτική και ουσιαστικά και κοινέ ε, κοινωνικές ε, ρήτρε και διατάξεις διότι σε σχέση με την ισοτιμία αυτού του ενιαίου νομίσματος ε, θα πρέπει να δούμε τη διαφορετική, τη διαφοροποιημένη θέση τώρα των κρατών που χρειαζόμαστε μηχανισμούς που θα ρυθμίζουν όλα αυτά. Κατά τούτο πιστεύω το σχέδιο και συμφωνώ απόλυτα με τον Άντριο Νταφ πρέπει να είναι φιλόδοξο, σοβαρό σχέδιο, με σοβαρή προσφορά που θα υποβάλουμε προς τους πολίτες. Να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται και γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι προοπτικές, οι φιλόδοξες προοπτικές και θα πρέπει να διαβουλευτούμε, να βρούμε δρόμους και δυνατότητες η οικονομική, δημοσιονομική, πολιτική κοινωνική ένωση να επιτευχθεί. Πώς θα τα καταφέρουμε και σε σχέση με την νομολογία του ε, συνταγματικού δικαστηρίου στη Γερμανία δεν είμαστε ομοσπονδιακό μόρφωμα Πώς λοιπόν ένα τέτοιο επικοδόμημα θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτούς τους ε, όρους και αυτούς τους στόχους. Πώς οι πολίτες μας ε, στα κράτη-μέλη θα μπορούν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και να συμμετάσχουν. Σε αυτά πρέπει να δώσει πιστικές απαντήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια και πιέζει λοιπόν ο χρόνος, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας ευχαρίστω θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή την εργασία, σε αυτό το έργο και αδειμονώ να δω πώς θα εξελιχθούν τα θέματα και οι συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στους δύο εισηγητές ε, να απαντήσουν. Ο Γκουαλτιέρη πρώτα. Θέλετε να απαντήσετε στην, στα σχόλια. Δεν μπορώ να απαντήσω σε λεπτομέρεια σε αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα που εφήγησαν εδώ. Πιστεύω ότι η συζήτηση που ήταν τόσο ενδιαφέρουσα δείχνει ότι χρειαζόμαστε πολύ χρόνο έτσι ώστε να συζητήσουμε αυτά τα σοβαρά θέματα. Και ελπίζω ότι το νέο έγγραφο εργασίας θα παράσχει τη βάση για αυτήν την σοβαρή συζήτηση. Όσον αφορά τα ζητήματα που έθιξε ο Άντριου, νομίζω το πρώτο σημείο η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να προσαρμοστεί σε διαφορετικό ε, ε, μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η δυνατότητα να προσαρμοστεί λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Από θεσμική άποψη, η... ο λόγος της καγκελαρίου Μέρκελ ήταν πραγματικά ένα βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με τα όσα μας είχε πει στην Μπρίζ. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, απόψεις ε, για την Ευρώπη. Η μία που θα βασίζεται μόνο στις συνθήκες και η άλλη που θα λαμβάνει υπόψη και τους πόρους. Εν πάση περιπτώσει όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία αυτά στην έκθεσή μας, δηλαδή και οπωσδήποτε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο αυτό το ε, πλαίσιο διακυβέρνησης. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αν αλλάξουν ή δεν αλλάξουν οι συνθήκες. Θα πρέπει να τα, πούμε αυτά στην έκθεση. Και τέλος, το ζήτημα της ενδεχόμενης αναθεώρησης ε, των συνθήκων ε, όσον αφορά την πολιτική γειτονία και όσον αφορά το ενδεχόμενο να εισαχθεί ένα νέο επίπεδο ε, σύνδεσης βεβαίως και αυτά θα πρέπει να συζητηθούν όλα όσον αφορά το περιφερειακό ζήτημα δεν ξέρω αμφιβάλλω λίγο διστάζω να το συμπεριλάβω γιατί νομίζω ότι είναι ένα άλλου είδους πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και φοβούμε μήπως ανοίξουμε και το κουτί της Πανδώρας που θα οδηγήσει σε άλλες ε, επιπτώσεις και περιπλοκές. Δεν το συζητήσαμε αυτό μέχρι τώρα γιατί είναι νέα πρόταση. Επίσης, για να απαντήσω στην ερώτηση, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα είναι ένα θέμα νομικής ε, υποχρέωσης. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες είναι δεσμευμένες, έχουν δεσμευτεί να ε, μπουν στο ευρώ και ε, χώρες οι οποίες έχουν σαφώς αποφασίσει να μην μπουν, που έχουν αποφασίσει το opting out. Η συνοχή της πολιτικής βούλησης βεβαίως σχετίζεται με, τη, με τους κύκλους τοπικής δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την νομική ε, βάση, το νομικό καθεστώς. Βεβαίως εξαρτάται και από τη δικιά μας ικανότητα να θεσμοθετήσουμε μια νέα διακυβέρνηση έτσι ώστε να μπορούμε να ξεπερνούμε τις ευρωκρίσεις ε, και έτσι ώστε η Ευρωζώνη να γίνει όχι μόνο οικονομικά ελκυστική αλλά και πολιτικά ελκυστική έτσι ώστε όλοι να θέλουν να γίνουν μέλη. Τέλος κύριε Σούλτς. Με μεγάλη προσοχή σας άκουσα. Ευχαριστώ αυτά, για αυτά που μας είπατε. Και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα συμμετάσχετε ενεργά στην συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ο Σέρχος Σταρκόφσκι θέλει να προσθέσει κάτι. Χαίρομαι γιατί δεν τα βλέπουμε τόσο άσχημα πια. Στο τελευταίο χαϊκού του Βαν Ρόμπουι με είχε απογοητεύσει. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι με το Ρομπέρτο μπορεί να συνεχιστεί τέτοια απεσιοδοξία. Και συμφωνώ με τον Ανδρέα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή. πριν την σύγκληση της συνέλευσης. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα μας πει και ο Βαν ή και αν θα είναι πιο επικοδομητικά αυτά που έχει να πει και δεν περιορίζονται στον εγωισμό του. Λοιπόν, από την έκθεση Βαντίντεμαν του 75 ακούγονται αυτά τα πράγματα 40 χρόνια δηλαδή σχεδόν και ξέρουμε που κατέληξαν. Στον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων στην Υγειά την Ιρλανδία. Ακούσαμε τα επιχειρήματα και τα υπέρ και τα κατά εκατοντάδες φορές. Το θέμα είναι θα υπάρξει καμία υποστήριξη στην ιδέα αυτήν. για τα πολυεπίπεδα στο κοινοβούλιο ξέρετε τι φρονώ. Πριν από έξι μήνες φαινόταν ότι δεν θα υποστηριχθεί η ιδέα αυτή στο κοινοβούλιο αλλά υποστηρίχθηκε και μεταξύ πολλών σημαντικών ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πολύ σωστό να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο ιδίως σε αυτήν τη φάση διότι το θέμα δεν είναι μόνο της εικόν αλλά του μέλλοντος του Κοινοβουλίου ολόκληρου. Συμφωνώ βέβαια με τον Ροβέρτο ότι πρέπει να σκεφτούμε και εκείνους που δεν αποκλείουν την πιθανότητα να μπουν μεν στην Ένωση αλλά και εμεί οι χώρες που είμαστε στην Ένωση δεν είμαστε στην Ευρωζώνη και άλλοι που θέλουν ίσως να σκεφτούν να μην μπουν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό ένα τέτοιο προηγούμενο και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερα διαδικαστικός. Για την σύνδεση ή για την συνδεδεμένη ένταξη που λένε associated membership. Οι χώρες που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται την ένταξη αλλά ξέρουμε ότι για να χρησιμοποιήσω έναν εμφημισμό ότι δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση και εννοώ την Τουρκία αυτή η ιδέα μιας έτσι βοηθητικής ένταξης ή associated membership ίσως είναι χρήσιμη. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι αυτό θα ενίσχυε την αξιοπιστία μας στα Μπαλκάνια. Υπάρχουν χώρες που τους έχουμε υποσχεθεί την ένταξη και πρέπει να πραγματοποιήσουμε την υπόσχεσή μας. Αν προτείνουμε αυτού του είδους την δευτερεύουσα ένταξη πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπονομεύει την αξιοπιστία του όλου σχεδίου. Ξέρω ότι ο Άντριου δεν το βλέπει έτσι αλλά θα μπορούσε να εκλειφθεί έτσι από την κοινή γνώμη γιατί η αναγνώριση των αδυναμιών μπορεί να εκλειφθεί ως αθέτηση υποσχέσεων ή και προς υποψήφιες χώρες και προς υπάρχουσες χώρες μέλη. Δεν πρέπει να παρετηθούμε τόσο γρήγορα γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις υποψήφιες αυτές χώρες και να κατακαιρματίσει την κοινή τους γνώμη. Εάν τελικά οι Βρετανοί αποφασίσουν ότι θέλουν να φύγουν από την Ένωση, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να το ενθαρρύνουμε κιόλα. Αν και μερικές φορές μας εκνευρίζει και άλλες φορές να μας σωθεί να τους το ζητήσουμε. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε πολύ τι εννοούμε, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες αυτές ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Γιατί μου φαίνεται ότι τελικά τελικά λέγω αν εμείς στην Επιτροπή μας δεν δείξουμε κάποια αισιοδοξία ποιος θα τη δείξει η όλη αυτή η ιδέα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σημαίνει ότι έχουμε ιδέες για τη μελλοντική λειτουργία της Ένωσης και πρέπει αυτό να το δείξουμε ρητά. Δεν είμαστε μόνο πολιτικοί αλλά και εμπειρογνώμονες εδώ στην Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά. πρέπει τελικά να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν είναι ανάγκη για να πετύχουμε τους στόχους μας να καταλήξουμε σε κατακαιρματισμό ή ολοκληρωτική ανασκευή όλων όσων λέγαμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τι θα πούμε. Παραδείγματος χάρη η ιδέα μιας υποεπιτροπής της εικόν ή της ε, δευτερεύουσας αυτής ένταξης μπορεί τελικά να ακουστεί σαν καταστροφική για τις ιδέες μας και να δώσει λάθος μηνύματα ότι δηλαδή αμυνόμαστε τώρα και δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να δείξουμε γιατί δεν τα λέμε αμυντικά όλα αυτά Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, και τους ε, δύο. Ελπίζω ότι μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε ένα έγγραφο εργασίας έτσι ώστε να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας γραπτό για να κάνουμε ακόμα πιο ενδελεχή συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγω. Ε, θα ζητήσω πάλι από την κυρία Λεγκρίπ να αναλάβει την Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια των εργασιών σας. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία αφορά την έκθεση του Προέδρου Κάρλο Καζίνη σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των αντιπροέδρων που εκλέγονται διαβοής. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2 που αφορά το άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο τμήμα της τροπολογίας 2 υπάρχει και προφορική τροπολογία κύριε Άνδρου Ντάφ ευχαριστώ πολύ το έχουν τα μέλη το έχουμε κυκλοφορήσει η προφορική τροπολογία θέλει να τροποποιήσει τον παρόντα ε, κανονισμό στο άρθρο 2 με τον, ε, ε, με τον κανόνα 13. που ζητάει αντιπροσώπευση των κρατών μελών. Είναι λίγο αρχαϊκή αυτή η διατύπωση. και απλώς νομίζω ότι θα πρέπει να εξευρεθεί η γεωγραφική ισορροπία που νομίζω ότι είναι μια πιο σύγχρονη διατύπωση. Κύριε Τασκόφση, το πρόβλημα είναι ότι η προφορική τροπολογία μόλις μας έχει η ε, υποβληθεί και ενδεχομένως αυτό το officers ε, ε, να είναι καλό στα αγγλικά αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Και έχω κι εγώ ένα πρόβλημα εδώ, έστω και αν υπάρχει γεωγραφική ισορροπία, δεν, με, δεν με ικανοποιεί και θα καταψηφίσω την τροπολογία αυτή. ο κύριος Ντάφα. Πα ότι με 27 χώρες μέλη είναι πολύ δύσκολο να εκπροσωπούνται όλες στο Προεδρείο από έναν βουλευτή. Αλλά δέχομαι ότι η προφορική τροπολογία απορρίπτεται. Δεν είναι αποδεκτή δηλαδή. Λοιπόν, η προφορική τροπολογία δεν θα ψηφιστεί, συμφωνούμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τώρα το πρώτο τμήμα της 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 2. Α, όχι, ναι. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται και αυτό. Επόμενη είναι δηλαδή 3, 4, 6, 7 δεν έχουν πια νόημα. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 5 υπέρ. Την 5 είπα. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Τώρα θα ψηφίσουμε την εξυπηρού Ρέγγελ γνωμοδότηση για τροποποίηση του κανονισμού εποπτείας κλπ. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Συμβιβαστική α, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα η συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 6 εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 8 περ κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές η εννέα εγκρίνεται τροπολογία 17 υπέρ κατά χες 17 εγκρίνεται 18 υπέρ κατά πόχες η 18 απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές η 19 απορρίπτεται συμβιβαστική γάμα υπέρ κατά χες εγκρίνεται Συμβιβαστική Δέλτα υπέρ. Κατά. Ποιες. Η συμβιβαστική Δέλτα εγκουρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται η 13. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εποχές. Η 1 εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. εποχές Η 14 εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κάτα. Οι η τρία εγκρίνεται τέσσερα περ κατά ψυχές η τέσσερα εγκρίνεται τώρα το σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα η έκθεση του κυρίου Νταφ Υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Πρώτα η 20 υπέρ. Κατά. Yes. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Ποχές. Η 21 εγκρίνεται. 89 υπέρ. Τα. Χες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ. κατά εποχές εγκρίνεται. Είναι 91 υπέρ αυτά. Ποχές. Τι είναι 91 εμπορίνεται. 23 υπέρ. αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 93

υπέρ κατά όχιες η 97 απορρίπτεται 98 υπέρ τα Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Τα. Χες. Εγκρίνεται 100 υπέρ. κατά Yes. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Yes. Εγκρίνεται 101 υπέρ. Α, κατά τμήματα, α, κατά τμήματα. Μάλιστα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ, της 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 26 υπέρ. κατά χες εγκρίνεται 102 υπέρ α χες απορρίπτεται 103 υπέρ κατά οχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές. Η 104 απαρρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Χες Απορρίπτεται 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 28 υπέρ. Τα χες εγκρίνεται 29 υπέρ τα χες εγκρίνεται 109 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Η 110 καταπίπτει. 111 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές η 117 εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. προχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Β υπά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα κατευθείαν η συμβιβαστική γάμα. Ορίστε κύριε Ντούφ. Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση εδώ πέρα που έχει διανεμηθεί που φέρνει πιο κοντά την πρόταση στη θέση της εικόνης στο στη συμβιβαστική πρόταση της εικόν. Λέει δηλαδή ότι η Προεδρία του Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο και θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μετά από σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να οργανώσει τη σχετική ακρόαση του υποψηφίου. Έχει κανείς αντίρρηση για αυτήν την προφορική τραπαλαγία. θα ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία του συναδέλφου μας Ανδρέου Νταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία αυτή, η προφορική, εγκρίνεται.

εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 128 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μας βλέπετε τους αριθμούς παρακαλώ. Για την 130-13 υπέρ, 9 κατά. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ 9 κατά 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Yes. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 134 ορισμένες πρόσθετες λέξεις. National Parliament of a Participating Country. Υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά απορρίπτεται 11-11 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά Χές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά Προχές. απορρίπτεται 141 υπέρ κατά Προχές. απορρίπτεται 142 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 143 υπέρ τα ποιες απορρίπτεται 144 υπέρ συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ο συμβιβασμός ε. 145 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 41 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 139. Μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό παρακαλώ. Λέει ο κύριος 10 υπέρ 11 κατά. 139 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 140, ε, 42 υπέρ Κατά. Ποιε. Απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Κατά. Ποιε. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά. αρχές απορρίπτωται. Σαράντα τρία υπέρ κατά αρχές απαρρίπτεται. Σαράντα υπέρ χεφ απορρίπτεται 45 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 46 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 47 υπέρ απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Τα. Χες. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ μετά Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκουρίνεται. Συμβιβαστική F ή σίγμα τάφη. Πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Ποιες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ζήτα ή Υπέρ. Κατά Εποχές. εγκρίνεται 58 υπέρ κατά Εποχές. απορρίπτεται 59 υπέρ κατά. Ποιες απορρίπτεται. εξήντα υπέρ κατά. Ποιες απορρίπτεται. Επτά υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Ο Χουτό υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Εγώ μέτρησα 11-11 λέει κάποιος. Καλά θα ξαναψηφίσουμε. Αλλά να ψηφίσετε όλες, ε. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε υπέρ απορρίπτεται. Εννέα. Εννέα. Γιατί οι προηγούμενες ήταν όλες μαζί. Τώρα 9 είπα, υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Α, όχι, όχι. 68. 68. 68. 68. Κατά. Εποχές εγκρίνεται δέκα υπέρ κατά χες εγκρίνεται εβδομήντα υπέρ κατά χες εγκρίνεται 71 71 λέγω υπέρ κατά χες απορρίψετε 11 υπέρ 11 κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ήττα υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. δεκατρία υπέρ. εγκρίνεται 14 είπε κατά εγκρίνεται Θέλετε το λόγο κύριε Γκουαλτιέρη, μάλιστα κυρία Πρόεδρε. Ζητώ για το γιοτά ψηφοφορία κατά τμήματα, το πρώτο και το δεύτερο. 34α χωριστά από το 34β δηλαδή. Α, εντάξει λοιπόν, κατά κατα τμηματα δεν υπάρχει αντίρρηση. Λοιπόν, για τη συμβιβαστική γιώτα το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Α. Χ. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα του συμβιβαστική γιώτα. Ποιος είναι υπέρ? Και contre. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές η τροπολογία 16 εγκρίνεται τροπολογία 67 υπέρ 77 συγγνώμη κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός J, κύριε Ντάφα. Για λόγους ε, συνεκτικότητας με αυτά που κάναμε στο συμβιβασμό C, οι λέξει elected, εκλεγμένος, που αναφέρεται την έκτη ε, αράδα πρέπει να τροποποιηθεί και να το να πούμε approved, όχι elected, approved. για λόγους εθυραμισμούς με τα όσα ήδη έχουμε ψηφίσει, θέτω σε ψηφοφορία το συμβιβασμό J, υπέρ. Και contre. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική τροπολογία απορρίπτεται. 10 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα λέει ο κύριος Νταφ. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 17 απερίφθη. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 81 εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 λέει αρχικά η Πρόεδρος. Όχι, μία προσθήκη. Μία προσθήκη, ε, ένα τμήμα της τροπολογίας 82. Ποιος ψηφίζει υπέρ αυτής της προσθήκης, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 87 υπέρ Contre <laughs> <laughs> <laughs> Qui s'abstient Αποχές. L'amendement est adopté. Εγκρίνεται η τροπολογία. Ωραία. Ψηφίζουμε επί του συνόλου της γνωμοδοτήσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. 18 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους. Συγχαρητήρια. Κύριε Μπρόκ, έχετε το λόγο. Κύριε Μπρόκ. Έχω ένα σημείο που έμεσα συνδέεται με αυτό. Ακριβώς τις συμβαστικές τροπολογίες μόλις τις διάβασα στην έκθεση Σιλβί στην Οικονομική Νομισματική Επιτροπή υποβάλλει κάποιες προτάσεις εδώ για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου σε όλα αυτά τα ζητήματα. Συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια που αντιβαίνει πλήρως στη μέχρι σήμερα θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι θεσμικό ζήτημα αυτό, σαφώς, και παρακαλώ να επανεξεταστεί αυτό. Αν η ΕΚΟΝ στα θέματα τα θεσμικά μπορεί να υποβάλει προτάσεις που δεν συνάδουν σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ή δεν είναι δική τους αρμοδιότητα. Ίσως η δεν ειναι δικη του αρμοδιοτητα μπορεί να το ελέγξει αυτό. Προτού ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή. Mr. Duff. Yes, Όπως πάντα, ο κύριος Μπρόκ έχει δίκιο. Και σαν εισηγητής θα μιλήσω με αυτούς που είναι υπεύθυνοι στην Επιτροπή ΕΚΟΝ σε μια προσπάθεια διευκρίνησης της θέσης του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Για να μην υπάρξει και προηγούμενο. Κύριε Γκολτιέρη, να προσθέσω ότι οτιδήποτε σχετίζεται με πιθανή τροποποίηση των συνθήκων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής, αλλά και ό,τι σχετίζεται με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο των θεσμικών της οργάνωσης αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Είναι επομένως απολύτως σαφές ότι ο συνάδελφος Μπρόκ έχει δίκιο όταν αναφέρεται στις δικαιοδοσίες της Επιτροπής εδώ συναγματικών υποθέσεων για να ε, συζητούν τέτοια θέματα. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο επ' αυτού. Όχι. Σημειώνουμε λοιπόν τις παρατηρήσεις ε, οι οποίες άλλωστε συγκλίνουν επί του θέματος αυτού και θα αποστείλουμε επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της Επιτροπής μας στην Επιτροπή ΕΚΟΝ αναφέροντας όλα αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε κι εσείς, ε, δηλαδή τις αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής Συναματικών Υποθέσεων ε, και θα δούμε τι μέλλον θα έχει, τι τύχη μάλλον θα έχει αυτή η επίσημη εντό εισαγωγικών επιστολή στον Πρόεδρο. Θα δούμε πώς θα συνεχίσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ακαμφόβες ζήτημα se faire jour ici au sein de notre euh, ε, μια και όλοι έχουν την ίδια άποψη στην Επιτροπή μας άλλωστε για το ζήτημα αυτό. Τελείωσε λοιπόν η ψηφοφορία και προχωράμε στο τελευταίο σημείο το οποίο είναι γεγραμμένο στην ημερήσια διάταξή μας. Πρόκειται για μία έκθεση του Προέδρου Κασίνη. Δεν είναι ακριβώς έκθεση, αλλά αφορά την ερμηνεία των άρθρων 186 και 187 του κανονισμού Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη σύνθεση των επιτροπών και του αναπληρωτές των εν λόγω επιτροπών. μια και απουσιάζει ο πρόεδρος Καζίνη, ο οποίος είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. δεν ξέρω εάν κάποια μέλη θέλουν οπωσδήποτε να συζητήσουμε σήμερα το θέμα, ε, γιατί εγώ θα ήθελα να προτείνω, μια και απουσιάζει ο πρόεδρος Καζίνη, ε, να ε, αναβάλουμε την ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος αυτού. Δεν ξέρω βέβαια αν κάποια ομάδα ή κάποιο μέλος θέλει οπωσδήποτε να παρουσιάσει κάποια σχόλια ή κάποιες παρατηρήσεις, αλλά βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψη του Προέδρου Καζίνη, δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε την άποψη δηλαδή, που έχει καταλήξει με τις εργασίες του ο κύριος Άντριου Ντάφα. Νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ε, επιστολή ως έχει χωρίς συζήτηση. Ε, γιατί δεν χρειαζόμαστε τον πρόεδρο Καζίνη. Υπάρχει η επιστολή του, υπάρχει η επεξήγηση. Κύριε Γκουαλτιέρη, θέλετε να, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας στηρίζει την πρόταση ερμηνείας των άρθρων 186 και 187 για τους λόγους για τους οποίους έχουμε ε, συζητήσει και έχουμε εξηγήσει και στην ε, ε, συζήτησή μας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αναλογική παρουσία των ε, μελών και στις επιτροπές έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα. Βάσει αυτών, λοιπόν, τον, αυτού του σκεπτικού μπορούμε να δεχτούμε την ερμηνεία που δίνεται στην επιστολή. Και εμεί συμφωνούμε με την ερμηνεία, επομένως μπορούμε να το ψηφίσουμε να περάσει αυτή η επιστολή. Ωραία. Λοιπόν, για να είμαστε πιο αποτελεσματικές και να λάβουμε υπόψη μας όλα τα αρμόδια κριτήρια όπως την απαρτία, αν θέλουμε σήμερα να εγκρίνουμε την ερμηνεία του Προέδρου Χασίνη και δεν διαφωνεί καμία ομάδα, τότε ας την εγκρίνουμε. Υπάρχει λοιπόν ομοφωνία εδώ να εγκριθεί η ερμηνεία του Προέδρου μας, μάλιστα θα υποβληθεί στον ίδιο. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, τελεία. Έληξε η συνεδρίαση.